Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Είμαστε πολλοί εδώ στην αίθουσα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την προσκεκλημένη μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου στο όνομα της Επιτροπής μας να καλωσορίσω την Πρωθυπουργό της ε, Σερβίας, ε, την κυρία Άννα Μπρεναπίτς. Καλώς ήρθες. Χαιρόμαστε πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω την ε, Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, την κυρία Γιατράγκα Γιοξίμοβιτς, που έρχεται τακτικά στις Βρυξέλλες, καθώς και την πρέσβυρα της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία Άννα Χρουστάνοβιτς. Καλώς ήρθατε. Βλέπετε ότι ε, είναι πολύ καλή η ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλλα εδώ. Ε, έχουμε μια αποκλειστικά ε, γυναικεία αντιπροσωπεία. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Ισταν Πάστορ βρίσκεται επίσης εδώ πέρα, όπως και ο πρόεδρος της κυβέρνησης Βορχοτίνα, ο κύριος Μύροβιτς. Είναι παρόν? Ωραία. και θα ήθελα να καλωσορίσω και ε, τον κύριο Σανφαπίτση, ε, ε, πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βελιγράδι. Όπως βλέπετε, το ενδιαφέρον για την επίσκεψή σας και για τη χώρα σας είναι μεγάλο. Κάποιες παρατηρήσεις από την πλευρά μου ως πρόεδρο της Επιτροπής αυτής, αλλά και ως εισηγητή για τη Σερβία. Από τον Ιούνιο είσαστε επικεφαλής ε, της σερβικής κυβέρνησης. Έχετε παρουσιάσει ένα φιλόδοξο θεματολόγιο εξυγχρονισμού. Βασίζεται στην ψηφιοποίηση, την καινοτομία και την εκπαίδευση. Υποσχεθήκατε να βελτιώσετε την δημοσιονομική εξυγίανση και να βελτιώσετε τις συνθήκες για την επιχειρηματικότητα καθώς και να δίνετε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, επαναλάβατε τη δέσμευσή σας ε, προς ε, Ανατολισμό, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με καλές ε, σχέσεις γειτονίας. Επίσης, στο τελικό του τη, μας δείξατε πόσο μπορεί να είναι κανείς πατριώτης χωρίς να είναι εθνικιστής. Ε, κυρία Πρωθυπουργέ, η, ε, η σε ένταξη της Σερβίας και του συνόλου των Δυτικών Βαλκανίων είναι κάτι που θα απαιτήσει χρόνο και προσπάθεια, αλλά ε, η απόδοση των, της επένδυσης, όπως το λέμε, αξίζει τον κόπο. Κύριε Πρωθυπουργέ, πέρα από την οικονομική ανάπτυξη της χώρας σας, θα θέλαμε να μας πείτε πώς βλέπετε την πολιτική κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Θέλουμε επίσης να ακούσουμε τα σχέδια σας όσον αφορά την ε, δημοκρατική ε, σταθεροποίηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, και την ελευθερία των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη χώρα σα μεταξύ άλλων θα πρέπει να δράτουμε κάθε ευκαιρία για να, έχουμε πραγματικό, να υπάρξει πραγματικός διάλογος ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα. Επίσης, ε, υποσχεθήκατε να εφαρμόσετε μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική πώς ε, συνδέεται αυτό με την υποχρέωση να ευθυγραμμίσετε την εξωτερική πολιτική της Σερβίας με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χωρίς πολλά λόγια σας δίνω το λόγο και θα δώσω το λόγο στους συναδέρφους για να σχολιάσουν αυτά που θα μας πείτε και να σας θέσουν ερωτήσεις. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much, David. Ευχαριστώ πολύ, David. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά όσο και τιμή να παρευρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας. Η νέα σερβική κυβέρνηση ανέλαβε πριν από 100 ημέρες περίπου και μεγάλη μου επιθυμία όσο και πρόθεση ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψή μου να είναι στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι ένα μήνυμα για το πού βαδίζει η Σερβία και πού θέλει να βρίσκεται. Thank, uh, Ευχαριστώ την πρεσβεία μας εδώ και όλους τους συναδέλφους μου αλλά και σας που καταστήσατε δυνατή αυτή την επίσκεψή μου. Βρίσκομαι εδώ με ιδιαίτερη χαρά ενώπιόν σας και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το προσωπικό μου όραμα για το μέλλον της Σερβίας. Το ερχόμενο Σάββατο, 14 Οκτωβρίου, θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω στους Σέρβους πολίτες τα αποτελέσματα των 100 πρώτων ημερών της διακυβέρνησής μας. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένη με τα όσα επιτύχαμε το πρώτο τρίμηνο, λίγο περισσότερο, τις πρώτες 100 μέρες της κυβέρνησής μας. Αρχίσαμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, ε, αντιμετωπίσαμε απεργίες αλλά αυτή τη στιγμή λύσαμε αυτά τα προβλήματα και δείξαμε ότι μπορούμε να εργαστούμε ως ομάδα, που είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου, προχωρήσαμε. Αυτή είναι η προτεραιότητά μου. Να δείξουμε ότι μπορούμε να εργαστούμε ως ομάδα και να προετοιμάσουμε τη Σερβία για ε, τη συντομότερη δυνατή ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρώτα απ' όλα και κυριότερα θα πρέπει να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν σκοπό να μας βοηθήσουν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να βελτιωθεί η κατάσταση στη Σερβία, να είναι καλύτερη η ζωή εκεί. Αφού αντιμετωπίσαμε λοιπόν τις απεργίες αυτές, βρεθήκαμε σε ένα έδαφος που είχαμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε την ε, καλή διακυβέρνηση του προκατόχου μου και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Αλεξάνδρ Βούζης. Τις επόμενες εβδομάδες μετά τις ε, απεργίες αυτές καταφέραμε να ε, έχουμε ένα επιτυχές πρώτο τρίμηνο 100 ημέρες. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το όραμά μου για τη Σερβία και τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και τον τρόπο με τον οποίο βλέπω εγώ τα πράγματα. Γιατί όταν αναλαμβάνεις πρωθυπουργό, αμέσως βρίσκεσαι σε μια θέση και μια κατάσταση που καλείσαι να επιλύεις τη μία κρίση μετά την άλλη και δεν έχεις χρόνο να προβληματιστείς, να σκεφτείς γενικότερα στρατηγικά το όραμά σου, που τι θέλεις να κάνεις για τη χώρα σου και που θέλεις να την οδηγήσεις, με ποιες προτεραιότητες. Θα σας πω λοιπόν πώς το βλέπω εγώ με την ιδιότητά μου. Όπως είπε ο Ντέιβιτ, μακάλιστε, η πρώτη και η δεύτερη προτεραιότητά μου στις προγραμματικές δηλώσεις ήταν τα εξής. Πρώτον, η ψηφιοποίηση και δεύτερον, η εκπαίδευση. Αν δούμε τη Σερβία ως ένα σπίτι, αυτό είναι ο θεμέλιος λίθος, η ψηφιοποίηση και η εκπαίδευση, η παιδεία. Η προηγούμενη κυβέρνηση έχει καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες για να αντιστρέψει την πορεία μας από τη χρεοκοπία. Πριν από τρία χρόνια η Σερβία πήγε τρεις μήνες από τη χρεοκοπία. Γι' αυτά τα λέει η Παγκόσμια Τράπεζα. Η προηγούμενη κυβέρνηση λοιπόν κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να ε, απομακρύνει αυτόν τον τιτανικό από το παγόβουνο. Έτσι ώστε η δική μας κυβέρνηση να έχουμε μια ισχυρή και στιβαρή βάση για την μελλοντική μας ανάπτυξη. Ευτυχώς εγώ ως νέος πρωθυπουργός δεν έχω να αντιμετωπίσω ε, μέτρα εξυγίασης οικονομικής και δημοσιονομικής που είναι πολύ ε, ε, αντιδημοφιλή και σκληρά. Ε, είμαστε στην επόμενη φάση. Πώς θα διαχειριστούμε τη δυναμική ανάπτυξη, τη βιώσιμη και την αϊφόρο για τη Σερβία. Αυτό μπορεί να γίνει με καλύτερη παιδεία, δηλαδή μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και ψηφιοποίηση. Για να γίνει αυτό, ιδιαίτερη ψηφιοποίηση, Έχουμε τεράστιο δυναμικό, τεράστιο ψηφιοποίηση. Δεν είναι μόνο περισσότεροι υπολογιστέ, αλλά ε, ψηφιοποίηση των διαφόρων κλάδων. Ε, μηχανοργάνωση ε, στις οικοδομές, στη γεωργία, στην υγεία, στην έρευνα, στην ανάπτυξη, ε, video games, δημιουργική κλάδι της οικονομίας, εκεί που ε, ανθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην Σερβία και όχι τώρα, τα τελευταία 5-6 χρόνια. Η ηλεκτρονική βιομηχανία στη Σερβία είναι εκείνη που αναπτύσσεται με τους ταχύτερους ρυθμούς, 10% ετησίως περίπου. Με ανάπτυξη λογισμικού που έχει ρυθμούς ανάπτυξη 20% ετησίως. Όλα αυτά που οφείλονται και από πού προέρχονται. Από νεοφυείς εταιρείε καινοτόμε, μικρομεσαίες, με λίγα λόγια. Αν αυτό λοιπόν συνέβη χωρίς καμία κρατική υποστήριξη, Αναρωτήθηκα, φανταστείτε τι μπορεί να γίνει με κάποια στοιχειώδη υποστήριξη από την κυβέρνηση. Άρα η ψηφιοποίηση και η παιδεία είναι τα θεμέλια πραγματικά για τη μελλοντική βιώσιμη αηφόρο και μακροχρόνια ανάπτυξη της Σερβίας. Αν χτίσουμε λοιπόν το σπίτι μας αυτά τα θεμέλια, έχουμε τρεις βασικούς πυλώνες. Οι τρεις βασικοί πυλώνες αυτοί είναι ακριβώς οι πυλώνες που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να προετοιμαστούμε για την ένταξή μας το συντομότερο στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια των Εθνών. Το πρώτο λοιπόν η οικονομική ανάπτυξη και μακροοικονομική σταθερότητα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ε, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και το τρίτο είναι το κράτος δικαίου. Αν σκεφτείτε αυτούς τους τρεις πυλώνες, γιατί ε, είπαμε ποια είναι τα θεμέλια και μετά ρίχνουμε τους τρεις βασικούς πυλώνες ε, του οίκου Σερβία, Στο πρώτο πυλώνα έχουμε προχωρήσει πολύ. Οικονομική ανάπτυξη και μακροοικονομική σταθερότητα. Όπω σα είπα, πριν από τρία χρόνια πήγαμε τρει μήνε από τη χρεοκοπία. Η προηγούμενη κυβέρνηση ενέκρινε και υλοποίησε ε, δέσμη μέτρων πάρα πολύ αντιδημοφιλή ε, εξυγίανσης δημοσιονομικής με δραστικές περικοπές των δημοσίων δαπανών. Σήμερα έχουμε 40.000 λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους σε σχέση με μια τριετία πριν. Χρειάστηκε να κάνουμε περικοπές 10% των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και στις συντάξεις επίσης. Και επίσης αναγκαστήκαμε να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τις δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυστηρούς ελέγχους των δαπανών για έργα υποδομών. Παρόλο που αυξήσαμε τις δαπάνες για έργα υποδομών, προσπαθήσαμε να γίνει αυτό στοχευμένα, με στόχο να ολοκληρώνονται τα έργα που είχαν αρχίσει. μάλλον να ολοκληρώνεται κάθε έργο που έχει ξεκινήσει πριν αρχίζουν ταυτόχρονα άλλα 100 και να μένουν όλα εμιτελή. Η σημερινή Σερβία λοιπόν κατάφερε να επιτύχει αυτή την εξηγίαση του προπολογισμού και τη μακροοικονομική σταθερότητα. Και εγώ κληρονόμησα μια κυβέρνηση με προϋπολογισμό τον καλύτερο προϋπολογισμό των τελευταίων 10 ετών. Το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό μας. Το δημόσιο χρέος άρχισε να μειώνεται, άρχισε να αναστρέφεται η τροχιά του και η πορεία του και στα τέλη του 2016 ήμασταν στο 73% του ΑΕΠ. Μιλώ για το δημόσιο χρέος. Σήμερα είμαστε γύρω στο 65%. Άρα συνεχίζουμε αυτή την καθοδική τάση. Αυτός ήταν ο βασικός πυλώνας όπου επιτεύχθησαν τα περισσότερα. Επίσης, είχαμε επιδόσεις στην ε, μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα και φυσικά χάρη στο νέο προϋπολογισμό και την υποστήριξη 80 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση με λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση για μένα είναι η απάντηση σε τρεις μεγάλες προκλήσεις. Το πρώτο είναι η διαφάνεια, ε, της δημόσιας διοίκησης. Το δεύτερο είναι η προβλεψιμότητα ε, της δημόσιας διοίκησης ως πολίτης, δηλαδή όταν απευθύνεσαι στο δημόσιο να ξέρεις τι απαιτείται από σένα, από έγγραφα να υποβάλεις και το τρίτο είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Γιατί αυτό είναι το θέμα, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Έχουμε ακόμα πολύ ε, δρόμο μπροστά μας. Και ο τρίτος πυλώνας είναι το κράτος δικαίου. Εμείς έχουμε επιδροθεί ιδιαίτερα στην εξηγένση του προπολογισμού, στον ισοσχελισμό του. Ε, δεν έχουμε επικεντρωθεί πολύ στον τρίτο πυλώνα. Αυτό είναι αυτό που μας περιμένει τώρα ιδιαίτερα τα κεφάλαια 23 και 24 πάρα πολύ βασικά για την ευρωπαϊκή μας ε, ολοκληρώση. Έρχομαι τώρα στη στέγη του σπιτιού. Η στέγη του οίκου Σερβία λοιπόν έχει να κάνει με την περιφερειακή σταθερότητα και κορονίδωλων αυτών η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περιφερειακή ε, σταθερότητα για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν μη τι άλλο, για λόγους εγωιστικούς τα τελευταία τρία χρόνια κάναμε πολλά έτσι ώστε η χώρα μας να σταθεροποιηθεί οικονομικά. Τώρα μπορούμε να δρέψουμε τους καρπούς από τη σταθερότητα αυτή, την φορολογική, τη δημοσιονομική, τη μακροοικονομική. Αλλά πώς θα δρέψεις καρπούς όταν είσαι σε μια περιοχή ασταθή. Ακόμα και αν η Σερβία είναι η μεγαλύτερη χώρα στην περιοχή μας, είμαστε αρκετά μικρή αγορά. Ε, οποιαδήποτε αστάθεια περιφερειακή μας επηρεάζει και μας. Αν υπάρχει αστάθεια στην περιοχή θα έρθουν λιγότεροι επενδυτές. Οι εμπορικές τράπεζες ή τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Παγκόσμια Τράπεζα κτλ θα σε δανείζουν πιο ακριβά γιατί θα πρέπει να συνυπολογίζουν αυτό το κίνδυνο. Άρα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας θα έχουν ακριβότερο δανεισμό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περιφερειακή σταθερότητα και ειλικρινά είμαστε βαθύτατα προσιλωμένοι σε αυτή. Η διαδικασία του Βερολίνου είναι βασικός φορέας περιφερειακής σταθερότητας και είμαστε βαθύτατα προσιλωμένοι στην διαδικασία αυτή του Βερολίνου. Και μετά, το επιστέγασμα είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όπως σας είπα και θα τελειώσω με αυτό. Η πρώτη φράση μου στις προγραμματικές δηλώσεις ήταν ότι ο στρατηγικός στόχος της Σερβίας είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θέλουμε να είμαστε μέλος στην ευρωπαϊκή οικογένεια των χωρών και των κρατών. τελευταία τριετία Ένα από τα πράγματα που μου άρεσαν και γι' αυτό αποφάσισα πέρσι τον Αύγουστο να μπω στην κυβέρνηση ήταν ότι η προηγούμενη σερβική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του τότε Πρωθυπουργού και νέου Προέδρου προώθησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ποτέ δεν είχε προβληθεί τόσο πολύ ε, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και δεν ακολούθησε το πιο εύκολο δρόμο, το λαϊκιστικό, ότι θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μας περιμένει ένα ε, κουβάς λεφτά στο τέλος του δρόμου. Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο η κυβέρνηση. Και εγώ εξακολουθώ να υποστηρίζω αυτό, ότι θέλουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές για μας τους ίδιους. Και δεύτερον, διότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που θα μας φέρουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομική σταθερότητα, ε, μεταρρύθμιση του δημοσίου για να είναι πιο αποτελεσματικό, πιο διαφανές, κράτος δικαίου, για να λειτουργεί καλύτερα η δικαιοσύνη και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Όλα αυτά είναι σημαντικά για τους Σέρβους πολίτες και για τις επιχειρήσεις μας. Άρα... Οι στόχοι αυτοί συμπίπτουν και ευθυγραμμίζονται. Εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες Θέσει εργασία για τους πολίτες. Ακόμα και αν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά, δεν πρόκειται η Ένωση να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για μας. Ούτε θα έχουμε άμεσα ωφέλη και ευημερία αυτόματη. Με αυτόν τον τρόπο προωθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διαφημίζουμε. Δεν θέλουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όσο ε, ο φτωχός συγγενής ε, που χρειάζεται βοήθεια και υποστήριξη. Και τη στιγμή που θα είμαστε έτοιμοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει τις θύρες να μας δεχτεί, θα είμαστε ένα ισότιμο μέλος, ίσο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι ο μόνος δρόμος για να προχωρήσουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Prime Minister. Εμείς ευχαριστούμε κυρία Πρωθυπουργέ και τώρα συνάδελφοι υπάρχει χρόνος για να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων έχουμε μέχρι τις 4 ώρες. Τέσσερις ακριβώς για μετά έχουμε το pre-fac να συζητήσουμε και έχει ανηλμένες προχωράσεις στις Βρυξέλλες για πρωθυπουργός. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κόκαν, ο οποίος είναι πρόεδρος της ε, Διακοινοβουλευτικής ε, Επιτροπής για Σταθεροποίηση και Σύνδεση. Δύο με τρία λεπτά σε παρακαλώ και κατώ μιλήσουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ βεβαίω. έτσι θα κάνω. Εξωγότατη κυρία Πρωθυπουργέ, καλώς ορίσατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας περιμέναμε πώς και πώς. Ε, έφτασαν τα, μαντάτα στις Βρυξέλλες ότι γίνεται Πρωθυπουργός ε, εκείνη τη μέρα ε, χαρήκαμε πάρα πολύ, θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά και για εσάς αυτό το γεγονός είναι ε, κάτι που σας ε, προσδίδει ευθύνε και ελπίζουμε επομένω να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Τώρα που σας άκουσα θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι είσαστε ε, ρεαλίστρια και ότι έχετε μια ούτως υπήν επιχειρηματική προσέγγιση επαγγελματική και μας είπατε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ότι είναι κορυφαία προτεραιότητα της χώρας πάρα πολύ σημαντικό να το ακούμε αυτό από τα χείλη σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ε, διαδικασία της περιφερειακής ολοκλήρωσης και υπάρχει καλή προϊστορία ε, αγαστών σχέσεων με την χώρα. Σχετικά πρόσφατα συνθήκαμε με τους ομολόγους μας από την σκούπιστηνα και ήταν πάρα πολύ θετική η συνάντηση αυτή και παραγωγική. Σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να μην παραβλέψετε το ποιοτικό στοιχείο σε κάποιες μεταρρυθμίσεις, όπως επίσης σε κάποιους τομείς που έχουν σχέση με την δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, καταπολέμηση της διαφθοράς, δημοκρατικών ελευθεριών, πολλές φορές ε, μας απασχολεί η κατάσταση των ΜΜΕ και η σχετική ελευθερία του τύπου είπαμε ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ούτως ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της ένταξης και βεβαίως θα απαιτηθούν συνταγματικές ε, αναθεωρήσεις. Οπότε είπαμε ότι ελπίζουμε να προτίθεται συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα περιπλοκά ζητήματα. Οπότε και πάλι να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας. Μπορείτε να υπολογίζετε στους φίλους που έχετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι το οποίο θα σας αναβαθμίσει τις φιλοδοξίες ούτως ώστε να αντεχθείτε στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια στο μέλλον και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Έντορτ, λέει ο πρόεδρος συνάδελφοι. Έχουν ζητήσει το λόγο αριθμός ρεκόρ 14. Άρα πρέπει έκαστος να πει κάτι, να κάνει την ερώτησή του, αλλά πει να αφήσουμε και στην κυρία Πρωθυπουργό ε, χρόνο απάντηση. Επομένω για τι 14 ερωτήσει πατρίε έχουμε 15 λεπτά. Επομένω, ένα λεπτό έκαστο πρώτο για το έργο κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρωθυπουργέ, καλώ ορίσατε. Σα εύχομαι καλό κουράγιο. Μ' ακούτε? Έλεγα καλώς ορίσατε και καλό κουράγιο για το έργο που έχετε αναλάβει. Σας ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Η πολιτική μας ομάδα, το Λαϊκό Κόμμα, υποστηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες της ε, Σερβίας για να βρει τον χώρο της στην Ευρώπη για ευημερία, ε, γιατί θα πρέπει να εξασφαλίζεται το κράτος δικαίου και η δημοκρατία. Έχω τρεις ερωτήσεις, ε, όπως είπαμε, για την ένταξή σας είναι ένας μαραθώνιος και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί η κοινή γνώμη θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος, καλύτερος φίλος της χώρας σας είναι η Ρωσία. Εσείς πώς θα τρέξετε σε αυτό τον ε, μαραθώνιο, θα σας ακολουθήσει αυτό το μαραθώνιο η κοινωνία. Ε, άλλη δεύτερη ερώτηση. Έχουμε ένα ψήφισμα πρόσφατα και λέμε στο σημείο υπαριθμό 26 ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί η νομοθεσία για τις μειονότητες. Ε, εσείς πώς αξιολογείτε την κατάσταση για την ρουμανική μειονότητα στην Σερβία. Τρίτον, δύο ε, λόγια για τον Άσαν Όριτς. Γιατί ε, έχουν δημιουργηθεί κάποιες εντάσεις για αυτό το θέμα με τις γειτονιάζουσες χώρες σας. Κύριε Πίτσουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας και καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σε συνέχεια τον ο κύριος ε, Πρέντα. Θα πρέπει να δούμε ε, αν σας εμπιστεύονται οι πολίτες σε αυτές τις προσπαθίες σας. θεωρεί ο κόσμος ότι η καλύτερη φίλη της χώρας είναι η Ρωσία και η Κίνα υπάρχει υποστήριξη σε αυτό το όραμα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Σε κάποια ε, γκάλοπ λένε τα δύο τρίτα των Σέρβων ότι δεν θέλουν ένταξη αν αυτό θα παραβλάψει σχέσεις με τη Ρωσία. Τι λέτε. Τι θέλετε να πείτε για αυτή την ε, κατάσταση έχετε ξεκινήσει αυτή τη διαδρομή του να κερδίσετε την κοινωνία. Ίσως ε, την υπόθεση ένταξη την παραβλάψει αυτή η κατάσταση. Α, όχι, δεν θα δεχόμαστε άλλους να ζητήσουν τον λόγο, λέει ο πρόεδρος. Λυπούμε. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο Τσουαλ Τάνοκ για το ΕΣΥΑΡ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αμπράνοπιτς, σας ε, Καλώς ορίζω θερμά. Θυμάμαι ότι σας είχα δεχτεί στο γραφείο μου με την προηγούμενη ιδιότητά σας ε, πριν κάποια χρόνια και ε, χαίρομαι πολύ που προχωρήσατε σε υψηλότερη θέση σε μια πολύ σημαντική χώρα των Δυτικών Βαλκανίων. Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες ε, και εμένα με ανησυχεί το γεγονός ότι σε αντίθεση με το Μαυροβούνιο για το οποίο είμαι εγώ εισηγητής και γι' αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η περιφέρεια αυτή Η χώρα αυτή προσχώρησε στο πακέτο των ε, κυρώσεων ε, κατά της ε, Ρωσίας λόγω της παρέμβασης στην Κρυμαία, ενώ εσείς όχι, κάτι που κατά τη γνώμη μου στέλνει λάθος μήνυμα όσον αφορά τις προσδοκίες σας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια αυτό είναι δική σας απόφαση και επικροτώ όλες τις ε, δέσμες ε, μέτρων ε, για τη μεταρρύθμιση που έχει οθετήσει η χώρα σας. Και τέλος ένα σύντομο μήνυμα προς εσάς. Εγώ προέρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και χαίρομαι που μπορώ... Ελπίζω σύντομα να δούμε να προσφορούν στην Ευρώπη όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Μην ακολουθήσετε το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου που μπορεί τότε να είναι εκτός. Ε, ευχαριστώ κύριος Βάιγκλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, εκφράσατε κάποιες πολύ σημαντικές σκέψεις σχετικά με τα κοινά συμφέροντα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να συνεργαστείτε μεταξύ σας ώστε να είσαστε ένα αξιόπιστο και σταθερό ε, μέρος της Ευρώπης. Θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για ε, κάποια αμφίσιμα σημεία της πολιτικής σας, ε, την Ρωσία και το Κωσυφοπαίδιο. δεν νομίζω όμως ότι η απάντηση σε αυτό θα είναι σύντομη. Η τελευταία μου ερώτηση. Εσείς ως Πρωθυπουργός πώς χειρίζεστε το πρόβλημα της ε, δημογραφικής αλλαγής. Είπατε ότι μειώσατε τις συντάξεις. Αυτό είναι καταστροφή για τους ηλικιωμένους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ήβος ε, από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι πολύ που έρχεστε τώρα για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες και αυτό ε, ελπίζω να ε, αποτελεί καλό ιονό και για το μέλλον, ε, να έρχεστε συχνά και στο μέλλον. Φυσικά όλοι ευχόμαστε να γίνετε σύντομα μέλος αυτής της οικογένειας. Ε, υπάρχουν όμως ακόμα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ε, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε πολλούς τομείς. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό ότι έχετε θέσει ως προτεραιότητα στην εκπαίδευση και την ψηφιοποίηση. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά θέματα, ε, έχετε επίσης μια καλή βάση για το μέλλον. Σημαντική όμως είναι και η περιφερειακή σταθερότητα και η σχέση με το γειτονικό κοσυφοπαίδιο, να υπάρχει διάλογος ε, και να γίνονται σεβαστές οι συμφωνίες και από τις δύο πλευρές. Μία σύντομη ερώτηση. αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνησή σας ε, και το περιβάλλον ε, και η ενεργειακή πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σπορκέζιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι Ιταλός Ευρωβουλευτής και δεν θα μπορούσα να αδιαφορήσω, δεν θα μπορούσα παρά να θέλω να έρθουμε πιο κοντά μια που είμαστε γείτονες και έχουμε και ιστορικούς λόγους να θέλουμε τις εξελίξεις αυτές. και για πολιτικούς λόγους και για πολιτιστικούς ε, αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας στο Βελγράδι και η σημερινή συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ σημαντική μια που στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θέλετε να κατοχυρώσετε και την ε, οικονομική, νομισματική σας ε, εθνική κυριαρχία. Σήμερα αυτή η κυριαρχία είναι η, το, δοθεμέλιο της ε, ελευθερίας. Τι λέτε. Ευχαριστούμε κύριε Μποργέσιο. Ο κύριος Επιτίδιος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ την ε, κυρία Πρωθυπουργό και εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της και στο έργο της χώρας της ε, στη διαδικασία εντάξεως της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία οπωσδήποτε υποστηρίζουμε. Ε, ήθελα να κάνω την εξή ερώτηση στα πλαίσια της προσελκύσεως επιχειρηματιών και επενδυτών ε, σήμερα επισκέφθηκε τη χώρα σας συνοδευόμενος από 150 περίπου επιχειρηματίες ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν. Ε, τι ακριβώς προσδοκάτε από την επαφή αυτή την επιχειρηματική με την Τουρκία. Δεδομένου ότι και η οικονομία της Τουρκίας δεν είναι σε ανθούσα κατάσταση αυτή τη στιγμή και από την άλλη πλευρά οι Τούρκοι όπου και αν έχουν εμπλακεί, έχουν εμπλακεί για να κυριαρχήσουν πολιτικά. Πώς αντιμετωπίσετε τον κίνδυνο της επεμβάσεως της ε, Τουρκίας στα πολιτικά θέματα της χώρας σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σούιτσα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, να σας πω, θα μιλήσω κρότικα. Στην παρουσίασή σας είπατε ότι η κυβέρνησή σας είναι προσανατολισμένη στην οικονομία και είπατε ότι είναι και τα θεμέλια αυτά η οικονομία. Δεν μιλήσατε όμως για τις σχέσεις σας με τη Ρωσία και έχουν σχέση και με την κοινή γνώμη και για τη γνώμη που έχει ο κόσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε ξεκάθαρα ότι είσαστε προσιλωμένοι στην ευρωπαϊκή πορεία και στην ένταξη της Σερβίας. Ούτε μιλήσατε καθόλου για το κοσυφοπαίδιο. Αναφερθήκατε στην περιφερειακή σταθερότητα χωρίς συγκεκριμένα παραδείγματα ε, για το Κόσοβο, ας πούμε. Και τώρα έρχομαι στην ερώτησή μου. Θα συνεχίσετε να εμποδίζεται το Κόσοβο να ενταχθεί στους διεθνείς οργανισμούς. Νομίζω θα ήταν ένα σαφές μήνυμα ότι επιθυμείτε την περιφερειακή σταθερότητα εάν συμφωνούσατε να ενταχθεί το Κόσοβο στους διεθνείς οργανισμούς. Ευχαριστώ. Κυρία Μούντι. Thank you. And, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Και χαίρομαι πολύ με την πολύ σπάνια εικόνα να έχουμε ένα πάνελ γεμάτο γυναίκες. Ε, καλώς ήρθατε. Μιλήσατε για την ε, ένταξη της ε, Σερβίας, ε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όμως πολύ σημαντικές ερωτήσεις κατά συνέπεια αυτού, για παράδειγμα. Το να εμφανίζονται σε επίσημες τελετές καταδικασμένοι άνθρωποι για εγκλήματα πολέμου. Και Υπάρχουν και ε, αρνητικές εκστρατείες ε, για ε, δημοσιογράφους που διερευνούν διάφορες υποθέσεις αντί να δίδεται μια αντικειμενική απάντηση σε αυτούς. Και έχουμε τον νέο διαμεσολαβητή και τον διορισμό του ενώ δεν έχει καμία εμπειρία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, ε, πώς ε, βλέπετε το θέμα του νέου αγωγού αερίου ανάμεσα ε, στη χώρα σας και την Κροατία. Από την άλλη, ο κ. Σιακόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο για αυτές τις πρώτες εκατομμύρες της κυβέρνησης. Συμφωνούμε σε αυτό που είπατε για κατάρτιση και για ψηφιοποίηση Επίση, θεωρούσα πάρα πολύ θετικό το ότι είσαστε υπέρ τη ελευθερία του τύπου και, τα των δικαιωμάτων τέλο πάντων των μειονοτήτων. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει σταθερότητα στην ε, περιοχή σας. Η Μπάνια Λούκα και το Βελιγράδι έχουν σχέσεις ισότητας γιατί είπαμε για τον Ντόντιτ ότι υπάρχει κάποια αντιπαλότητα. Ο Βούτσιτς ε, είπαμε ότι μπορεί να πει στον ε, Ντόντικ ε, αρκετά. Εσείς. Thank you. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ζόφκο. Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, καλώς ορίσατε, συγχαρητήρια για αυτές τις επιτυχίες των πρώτων 100 ημερών της κυβέρνησης. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συναδέλφοι που μας μίλησαν για την περιφερειακή σταθερότητα. Συμφωνώ με το όσο είπε ο κύριος Πρέντος και ο δισηγητής μας. Η Σερβία και η Κροατία θα πρέπει να διαδραματίζουν επικοδομητικό ρόλο, να λυθούν έτσι τα προβλήματα της Βοσνίας και Ερσεγοβίνης. Υπάρχουν τώρα προβλήματα εκεί σε σχέση με το εκλογικό δίκαιο Οπότε για πέστε μας, ε, τι λέτε, τι μπορεί να κάνετε στο μέλλον, ούτως ώστε και η Βοσνία να έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Αν υπάρχει αστάθεια στην Βοσνία, θα υπάρχει αστάθεια και στη Σερβία. Αλλά θα πρέπει να ασχοληθείτε πιο εντατικά με τα προβλήματα στην ε, Βοσνία. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρος, και τώρα. Ο κύριος Μποστινάρου έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, κυρία Άννα Μπερνάμπιτση, αν το προσφέρω εδώ το όνομά σας, μεγάλη μας χαρά σας υποδεχόμαστε και πρώτα πρώτα ως Ρουμάνος δεν θα μπορούσα να χάσω την ευκαιρία να σας υποδεχτώ, αλλά ως σοσιαλιστής πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτική μας ομάδα θέλει την διεύρυνση προς τις χώρες των Βαλκανίων. Πρώτα πρώτα, για να δούμε τη διεθνή συγκυρία στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν έχουμε μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση που εμπλέκεται στην ε, περιοχή. Υπάρχουν και άλλοι. Και πολλές φορές τα θεματολόγια, τα συμφέροντα ε, είναι απλώς αποκλίνοντα. είναι και αντίθετα. Οπότε έχουμε σαν πρόσφατες εξελίξεις ε, και θετικές είναι το ότι πήγε στη Βάρνα ο κύριος ε, Βούτσης και σε συνεννόηση με Βουλγάρους και Έλληνες ε, συζήτησαν βλέποντας πάρα πολύ την ε, διεύρυνση και αυτό έχει σχέση με την επερχόμενη βουλγαρική και ρουμανική προεδρίας. Οπότε εσείς προτίθεστε να ευθυγραμμίσετε την εξωτερική σας πολιτική με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της άμυνας. Σε αυτή την περίπτωση θα έχετε πάρα πολλούς υποστηρικτές εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα κύριο Ζηλμούβιτς για την Άλτα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ό,τι καλύτερο εύχομαι στην χώρα, στην ευρωπαϊκή της διαδρομή. Ελπίζω σύντομα να πετύχετε αυτό το οποίο θέλετε. Νομίζω ότι τα πάτε πάρα πολύ καλά Τώρα ε, ερώτηση σε σχέση με την περιφερειακή σταθερότητα. Τι μπορεί να κάνει η χώρα σας ούτως ώστε να κάμψετε τις αποσχιστικές τάσεις στην Βοσνία. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε να έχει σταθερότητα η Βοσνία, γιατί αυτό είναι κάτι που το χρειάζεται και η δική σας χώρα εκτός από τη Βοσνία και χρειάζεται και για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γκάλα. Κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε Πρωθυπουργέ και από πλευρά μου. Ερωτώ. Αυτή η διαδρομή σας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι ε, ανεπιστρεπτή και τι γίνεται με την κοινωνία σας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σας την ευλογεί αυτή την πορεία. Γιατί υπάρχουν κάποιες φωνές ε, που ε, συγκαλυμμένα ή ανοιχτά ε, υποστηρίζουν στην Πάνια Λούκα τον Ντόντικ που θέλει να κάνει ένα δεύτερο δημοψήφισμα να κηρύξει ανεξαρτησία και να άξει στον αέρα τη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Εσείς επίσημα είστε κατά του βήματος αυτού. Η Κροατία είναι προνομιούχος εταίρος στο δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. όχι μόνο επειδή είναι πολύ κοντά σας η γλώσσα, γιατί μπορεί να διαβάσετε και όλα τα έγγραφα ε, στα κροατικά, αλλά ε, μήπως και ως ένα στοιχείο συμφιλίωσης που χρειάζεται ακόμα ε, μετά από όσα έγιναν πριν από λίγες δεκαετίες. Ευχαριστώ. Τελευταίοι δύο μιλητές από τη Σλοβενία, ο κύριος Πέτερλε πρώτος. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ, που είχε την καλοσύνη να αναφερθεί στο τελικό του Eurobasket και ξέρετε ότι ο σπόνσορας των ε, Σέρβων ήταν Σλοβαίνος και των Σλοβαίνων Σέρβος. Ιδού λοιπόν, οποία εταιρική σχέση και συνεργασία. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρωθυπουργέ για τα λόγια σας, πολύ σταράτα και πολύ ρεαλιστικά και συγχαρητήρια για τις πρώτες 100 μέρες. Χαίρομαι ε, για τη συνέχεια που έχει η κυβέρνηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων και της Ευρώπης που ε, άρχισε ο Πρωθυπουργός Βούτσης τότε και χαίρομαι που συνδέεται τη μακροοικονομική σταθερότητα με το κράτος δικαίου. Αν δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου, δεν νοείται πραγματική ε, κοινωνική οικονομία της αγοράς. Συμφωνώ με τα όσα είπατε και για την περιφερειακή σταθερότητα. Και άλλη μια ερώτηση, ε, εκτός των άλλων που έγιναν. Τι σκοπεύετε να ε, κάνετε σε σχέση με τη Βοσνία, η Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πεπισμένος ότι η Σερβία είναι όρημη για να διαπραγματευτεί νέα κεφάλαια και καλή επιτυχία σας εύχομαι και χωρίς καθυστερήσεις. Ο Φρανς Πόκοβιτς, ενεργός φίλος της Σερβίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλώς κύρια Πρωθυπουργέ. Ε, Καλωσορίζω και την Υπουργό και την Πρέσβη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγχαρητήρια για τις ε, πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησής σας και ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Μας παρουσιάσετε το δρόμο των μεταρρυθμίσεων που έχει πάρει η Σερβία και είναι πραγματικά ο μονόδρομος αν θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πιστεύω ότι ειλικρινά το επιθυμείτε. Εγώ θα πρέπει να μιλήσω και ε, για το Ευρωμπάσκετ, αλίμονο. Ε, συγχαρητήρια και συγχαρητήρια και για την εικόνα που δώσατε με τον ε, πρόεδρο της Σλοβενίας, Τσέρα. Ε, συγχαρητήρια που δείξατε ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε στην περιφέρεια μας. Δύο λόγια τώρα για τα υπόλοιπα. Τι θα κάνετε με τη δημογραφική πρόκληση. Οι γεννήσεις μειώνονται και ο κόσμος φεύγει από τη Σερβία. Τι θα κάνετε για να αποφύγετε τα προβλήματα της δημογραφικής αλλαγής, έτσι ώστε οι διάφορες περιφέρειες στην ε, Σερβία να αναπτύσσονται εξίσου, να μην είναι όλα στο Βελιγράδι. Πολλές ερωτήσεις έγιναν. Πρωθυπουργέ, βλέπετε το μεγάλο ενδιαφέρον ε, που έχει η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις στη χώρα σας. Τώρα έχετε το καθήκον να τα συνοψίσετε όλα αυτά μέσα σε 12 το πολύ 15 λεπτά. Και ε, τότε να αρχίσω αμέσω. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και το ενδιαφέρον σας. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες. Ζητώ συγγνώμη εάν ξεχάσω κάτι. Θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω όλα. Έγιναν πολλές ερωτήσεις, οι περισσότερες για τη σχέση μας με τη Ρωσία και σε κάποιο βαθμό και με την Κίνα. Θα ήθελα να σας πω το εξής. υπουργό Υπουργός Γιωξίμοβιτς και το Υπουργείο της ε, βολιδοσκοπούν συχνά την κοινή γνώμη σε δημοσκοπήσεις. Και από ό,τι είδαμε, σήμερα μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές οι δημοσκοπήσεις, «41% ήταν πέρσι και φέτος 49% ενώ συνολικά 66% ε, το 100 είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Και για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής και ο μεγαλύτερος υποστηρικτής και το ε, αντιλαμβάνεται και ο κόσμος αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ε, και κατά την άποψή μου αλλάζει η εικόνα ε, του κόσμου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργά αλλά σταθερά. Και προσωπικά θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω και να προωθήσω την υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο με προενταξιακά κονδύλια, αλλά με συνεργασία στην έρευνα, την ανάπτυξη, σε έργα υποδομών ε, που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κτλ. Also tell you Για να σας πω την αλήθεια, όταν είδα αυτό ότι τα δύο τρίτα των Σέρβων δεν είναι υπέρ της Ευρώπης, μα δεν είναι δυνατό να είναι σωστό αυτό. Γιατί αν δείτε τη Σερβική Βουλή, το 80% περίπου των βουλευτών μας προέρχονται από, δύσκολα, από διαφορετικά πολιτικά κόμματα Βέβαια, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα που έχει την πλειοψηφία ε, ε, έχει σχηματίσει και την κυβέρνηση, είναι σαφώς υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ε, ορισμένα από αυτά είναι υπέρ της Ευρώπης. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια εθνικιστικά δεξιά κόμματα, αλλά αυτά είναι μειοψηφία. Δεν μπορείτε να πείτε ότι τα δύο τρίτα του κόσμου είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ τα πολιτικά κόμματα κατά 80% στο Κοινοβούλιο να είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι πάει στραβά εκεί, αν το σκεφτούμε. Τουλάχιστον 49% λοιπόν ε, των πολιτών υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η Ένωση ως μεγαλύτερος υποστηριχτής και δωρητής. Η σχέση με τη Ρωσία. Προφανώς η σχέση με τη Ρωσία είναι κάτι το οποίο δεν κρύβει η Ρωσία. Έχουμε παραδοσιακά καλές σχέσεις, δεν κρύβει η Σερβία, συγγνώμη, με τη Ρωσία. Έχουμε πολιτιστικούς δεσμούς, θρησκευτικούς, προφανώς. Πολλοί Σέρβοι θεωρούν τη Σερβία φίλο. Γιατί μας υποστήριξαν στη δεκαετία του 90, γιατί αντιστάθηκαν ε, στον βομβαρδισμό της Σερβίας από τον ΝΑΤΟ για όλους αυτούς τους λόγους. Αλλά επίσης και σημαντικά έχουμε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Ρωσία. Είναι σημαντικό αυτό για την οικονομία μας. Και επίσης είμαστε εξαρτημένοι από τις αγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Έχουμε λοιπόν αυτή τη θέση με τη Ρωσία που δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αυτό ε, επηρεάζει, επεμβαίνει στη στρατηγική μας προσέγγιση για την ε, ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα και η δική σας χώρα, οι δικές σας χώρες συνεργάζονται με τη Ρωσία, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αλλά από τότε που ανέλαβα, ε, πρωθυπουργός, έχω ε, κοιτάξει διάφορα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκπληκτικό η αντίληψη που έχει ο κόσμος για τα πράγματα. Εσείς ως Ευρωβουλευτές θα πρέπει να συζητάτε θέματα με βάση τα γεγονότα και όχι την αντίληψη και το κλίμα που δημιουργείται. Και όταν λέτε ότι η Σερβία, για παράδειγμα, στρατιωτικά είναι πιο κοντά στη Ρωσία, θα ήθελα να σας πω ότι το 2016, δεν το λέω γιατί και εγώ εξεπλάγει. Το 2016 η Σερβία συνολικά είχε 16 πολυεθνικές ασκήσεις στρατιωτικές διαφόρων τύπων, 16. 9 από τις οποίες ήταν διμερείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 με τη Ρωσία, 2 με άλλες χώρες των Βαλκανίων, 2 με το ΝΑΤΟ μέσω της εταιρική σχέση για την ειρήνη και μία άσκηση με την Ουγγαρία. Το 2017 η Σερβία, σήμερα δηλαδή, συμμετείχε σε 13 στρατιωτικές ασκήσεις διακλαδικές, όπου μάλλον διορθώνει η Πρωθυπουργό, 13 με τον ΝΑΤΟ από 15, 7 διμερείς με τις Ηνωμένε Πολιτείε, 2 με τη Ρωσία από τις 15. Αυτή είναι η αριθμή και τα στοιχεία. Και είναι πολύ διαφορετική από την αίσθηση που έχει ο κόσμος. Αλλά όλοι έχουμε συνηθίσει να ακούμε ότι η Σερβία και η Ρωσία και τα λοιπά. Αλλά ας δούμε τους αριθμούς. Ο κύριος Τάνοκ μίλησε για την επιθυμία για την ευρωατλαντική μας ένταξη. Είμαστε σαφέστατοι και το λέμε ειλικρινά και ξεκάθαρα. Δεν θέλουμε ευρωατλαντική ένταξη. Θέλουμε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να γίνουμε μέλη του ΝΑΤΟ. Θέλουμε να διατηρήσουμε τη στρατιωτική μας ουδετερότητα. Αλλά αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι είμαστε ειλικρινά ουδέτεροι στρατιωτικά. Για να μην πω ότι συνεργαζόμαστε περισσότερο με το ΝΑΤΟ μέσω της ε, εταιρικής σχέσης για την ειρήνη, Partnership for Peace. Συνεχίζω. Εθνικές μειονότητες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό για τη Σερβία. Αλλά δεν μπορείτε παρά να αναγνωρίσετε ότι η Σερβία στην Ευρώπη είναι από τους πρωταθλητές στο σεβασμό των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων. Ακόμα και μετά την αιματηρή δεκαετία του 90, σήμερα η Σερβία είναι εκείνη η χώρα η οποία έχει τις περισσότερες εθνικές μειονότητες. 26 επίσημες, 26. Όλες αναγνωρισμένες ως εθνικές μειονότητες. Και έχουμε και το θεσμό των Συμβουλίων Εθνικών Μειονοτήτων έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική ζωή της Σερβίας. 21 τέτοια συμβούλια έχουμε, τα οποία συνεργάζονται ε, στο Συμβούλιο όπου προεδρεύει η Πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα. Προείδρευσα σε ένα τέτοιο ε, συμβούλιο. 15 διαφορετικές γλώσσες έχουμε στα σχολεία, στην εκπαίδευση στη Σερβία. Σε 15 διαφορετικές γλώσσες. Έχουμε 6 διαφορετικές επίσημες γλώσσες σε διάφορους δήμους, ιδιαίτερα στη Βόηβοντίνα. Άρα δεν μπορείτε να λέτε και στη Σλοβενία για παράδειγμα μέγας φίλος μας, αλλά οι Σέρβοι δεν θεωρούνται εθνική μειονότητα, δεν αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Και ούτε καν το ανοίγουμε αυτό το θέμα. Οι Ιταλοί αναγνωρίζονται, οι Ούγγροι, οι Σέρβοι όχι. Παρόλο που οι Σέρβοι είναι η μεγαλύτερη εθνική μειονότητα στη Σλοβενία. Άρα, σας παρακαλώ, για το θέμα των εθνικών μειονοτήτων, πιστεύω ότι η Σερβία κάνει πολλά πράγματα, είναι πολύ σημαντικό για μας και για να είμαι ειλικρινής είμαι πάρα πολύ περήφανη για τα όσα πράττουμε για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εθνικών μειονοτήτων. Περικοπές στις συντάξεις, βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας και πάντα είναι ένα θέμα συζήτησης. Αυτό που ρώτησε ο κύριος Βάγκελ. Κύριε Βάγγελ, ήταν απαραίτητο διότι πριν τις εκλογές, πριν την προηγούμενη κυβέρνηση, το 2012-2013 ανέλαβε η κυβέρνηση αυτή, είχαν αυξηθεί οι συντάξεις με πολιτικές αποφάσεις, με τρόπο μη βιώσιμο. Χρειάστηκε να κάνουμε περικοπές για να μπορούμε να τις πληρώνουμε τις συντάξεις χωρίς να χρεοκοπήσει η χώρα. Έκτοτε όμως, ακριβώς λόγω των μέτρων εξυγίανσης του προϋπολογισμού, αυξήσαμε δύο φορές τις συντάξεις. Όχι πάρα πολύ, πλην αυξήθηκαν. Όσο μπορούσαμε και σήμερα σκεφτόμαστε να αυξήσουμε αρκετά τις συντάξεις και το Οκτώβριο, στις 13 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις ε, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ελπίζω ότι το Σάββατο να έχω την ευκαιρία να το ανακοινώσω. Για πρώτη φορά λοιπόν θα έχουμε υψηλότερες συντάξεις στη Σερβία από ότι πριν το 2013 της κρίσης. Υψηλότερες συντάξεις. Αλλά τώρα σε γερά θεμέλια και σταθερά. Όπως και για τους μισθούς. Για τους εργαζομένους στην υγεία και στην παιδεία. Για πρώτη φορά τώρα μετά την τελική αύξηση που ελπίζω να ανακοινώσω την, ε, το Σάββατο, θα είναι ψηλότερη μισθή για πρώτη φορά μετά την κρίση, αλλά για πρώτη φορά σε υγιή βάση. Κόσοβο. Και περιφερειακή συνεργασία. Το κοσυφοπαίδιο. Είναι για τη Σερβία εξαιρετικά σημαντικό, αλλά θέλω να σας θυμίσω. Πριν από 4,5 χρόνια υπογράψαμε τη Συμφωνία των Βρυξελών. 4,5 χρόνια. Η συμφωνία των Βρυξελών ήταν πάρα πολύ σκληρή να υπογραφεί πολιτικά. Ήταν πολύ δύσκολη και υπεύθυνη απόφαση για να την πάρουμε. Ακόμα και σήμερα, ακόμα και στην τελευταία προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές, για τον κύριο Βούτζης, τον κατηγόρησαν τα δεξιά κόμματα και τα υποτιθέμενα ε, δημοκρατικά και υποψήφοι ότι υπέγραψε τη Συμφωνία των Βρυξελών και ξεπούλησε το Κόσοβο. Η Σερβία ε, τα έχει υλοποιήσει τα περισσότερα, αλλά η ραχοκοκαλιά της συμφωνίας είναι ε, ε, η ίδρυση της κοινότητας των σερβικών δήμων και κοινοτήτων. Και ούτε κατά διάνοια δεν έχουν αρχίσει να το εφαρμόζουν αυτό. Παρακαλώ, κοιτάξτε ποιος εφαρμόζει τη Συμφωνία των Βρυξελών. Ζητούν ακόμα από τη Σερβία, θα κάνετε το α, το β, θα τους πλογκάρετε στους διεθνείς οργανισμούς. Η Πρίστινα δεν υλοποιεί την ίδια την ουσία τη ραχοκοκαλιά της Συμφωνίας των Βρυξελών. Ο πρόεδρος ζήτησε να γίνει διάλογος για το Κόσοβο και αυτό πραγματικά είναι ένα σημείο ε, πολιτικής και ένα μήνυμα υπεύθυνης πολιτικής και γενναίας όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, η κοινωνία των πολιτών, οι οργανώσεις συμμετέχουν, ε, η εκκλησία, τα μίντια, άλλες ε, θρησκευτικές ενώσεις, όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει για να πει ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο μέλλον του πεδίου. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες για τις συνέπειες. Αυτό είναι πραγματικά μια γενναία στάση και πιστεύω ότι θα μας δώσει και μια ένδειξη για το μέλλον και τι μπορεί αυτό να σημαίνει και να φέρει. Αλλά πραγματικά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Σερβία έχει δείξει υπεύθυνη στάση. Ειλικρινά η Πρίστινα όχι. Η περιφερειακή σταθερότητα στη Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Ξανά και ξανά λέμε και επαναλαμβάνουμε ότι η Σερβία είναι εγγυήτρια δύναμη στη συμφωνία του Ντέιτον. Ότι χρειαζόμαστε τη Βοσνία Ζεγοβίνη ως χώρα, όπως έχει σήμερα. Και βέβαια έχουμε στενούς δεσμούς με τη Ρεπούμπλικα Σέρβσκα και προφανώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υποστηρίζουμε τη Βοσνία Ζεγοβίνη ως μία ενιαία χώρα με τη μορφή που έχει σήμερα. Η πρώτη επίσκεψη του Προέδρου Βούτσιτς ήταν στο Σαραγεύο. Μέχρι τα τέλη του έτους θα συνεδριάσουμε μαζί με την κυβέρνηση της Βοσνίας Σερζεγοβίνης, και με χαρά να συνεργαστούμε και να λύσουμε όλα τα εκρεμή ζητήματα. Και επ' ευκαιρία θέλω να σας πω ναι, ότι η Σερβία είναι εγκύτρια δύναμη της συμφωνίας του Ντέιτον. είναι μια αναστρέψιμη πορεία της ε, Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Κατά την άποψή μου είναι. Αλλά τι να σας πω. Πάντα έχουμε θέματα περιφερειακής σταθερότητας. Εξημότιμος βουλευτής με ρώτησε για την υπόθεση Νάσερ Όριτς. Αυτά είναι πράγματα που πληγώνουν βαθιά την περιφερειακή σταθερότητα. Εμείς είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι και ενοχλημένοι. Δεν φταίει κανείς, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν φταίει κανείς για τις φαγές ε, των Σέρβων πολιτών αμάχων στη Βοσνία. Δεν φταίει ο Νασερόριτς. Ποιος φταίει, κανένας άλλος και αυτό πληγώνει την περιφερειακή σταθερότητα. Διότι πραγματικά εμείς είμαστε προσιλωμένοι στην σταθερότητα της περιοχής μας και παραμένουμε ε, και ευέλικτοι και ανεκτικοί και ανοιχτοί στην επικοινωνία μαζί τους. Προφανώς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, αλλά σας παρακαλώ θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί και να πούμε ότι κάποιος θα πρέπει να ε, είναι υπεύθυνο για τον πόλεμο. Έγινε μια ερώτηση για καταδικασμένους για κλίματα πολέμου που εμφανίζονται σε δημόσιες τελετές. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαν στη Χάγη, παρα, τους παρέδωσαν οι... κυρίως η Σερβική Δημοκρατία ή παραδόθηκαν οι ίδιοι οικειοθελώς, δεν ξέρω τι και να έγινε, δικάστηκαν, καταδικάστηκαν, εξέτησαν την ποινή τους απελευθερώθηκαν και επέστρεψαν στη Σερβία. Δεν είναι επίσημοι, δεν είναι κυβερνητικά στελέχη, δεν είναι σύμβουλοι της κυβέρνησης. Είναι ελεύθεροι άνθρωποι, πολίτες. Υπάρχουν και άλλες χώρες στην περιοχή με εγκληματίε πολέμου που είναι στην κυβέρνηση και έχουν επίσημες θέσεις. What, what, you know, what... Άρα τι θα τους κάνουμε αυτούς. Ε, εξέτησαν την ποινή του. φυλακίστηκαν, απελευθερώθηκαν, επέστρεψαν. Δεν έχουν δημόσια αξιώματα. Πάντως και πάλι διαφέρουν οι καταστάσεις στην περιοχή μας. Και αυτό ε, διασαλεύει την περιφερειακή σταθερότητα. Εγώ είμαι δεσμευμένη και προσιλωμένη να συνεργαστώ με τους πάντες για να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Ενέργεια και περιβάλλον έχω χρόνο. Ε, ρώτησε ο Ιγκορ Σόλτες. Και πάλι δύο θέματα. Πρέπει να λέμε ξεκάθαρα ότι η νέα κυβέρνηση είναι φιλοευρωπαϊκή. Ακρεφνώς. Είναι πρώτη προτεραιότητα. Έχουμε δύο νέα υπουργεία στην κυβέρνησή μας. Το ένα είναι Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Και έχουμε και Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος. Προηγουμένως αυτό εντασσόταν στο Υπουργείο Γεωργίας. Τώρα δημιουργήθηκε ξεχωριστό Υπουργείο γιατί ξέρουμε ότι θα είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και από τα πιο δύσκολα και πιο δαπανηρά κεφάλαια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε Υπουργείο ξεχωριστό και είμαστε ακριβώς προσιλωμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Το ενεργειακό. Ξέρετε ότι Αρχίσαμε μεγάλα έργα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προσπαθούμε να έχουμε όλο και περισσότερη διαφοροποίηση στο ενεργειακό μας μείγμα και ένα βασικό έργο προτεραιότητας ήταν ο, ο αγωγός διασύνδεσης ε, για το φυσικό αέριο μεταξύ Βουλγαρίας και Σερβίας. Είναι πολύ σημαντικό για τη διαφοροποίηση στον ανεφοδιασμό και την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκα με τον Υπουργό Ενέργειας για να δω που βρισκόμαστε σε αυτό το έργο. I think... Ε, ε, σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι προσπάθησα να απαντήσω. Α, ερευνητική δημοσιογραφία, πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να είμαι ειλικρινής εδώ, ειλικρινέστατη και ανοιχτή για τη συζήτηση. Το έχω πει και στους δικούς μας δημοσιογράφους και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Σερβία, το λέω και σε εσά. Εγώ δεν καταλαβαίνω το θέμα αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Τι πρόβλημα υπάρχει, δεν έχουμε ερευνητική δημοσιογραφία στη Σερβία. Μπορεί να υπάρχει έλλειψη, αλλά όχι επειδή την καταστέλει η κυβέρνηση, αλλά επειδή δεν υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία στη Σερβία. Είναι πολύ λίγη η αντικειμενική. Είτε κάποιος είναι ακρεφνός φιλοκυβερνητικός ή ακρεφνός κατά της κυβέρνησης. Πολύ σπάνια είναι αντικειμενική η δημοσιογραφία. Υπάρχουν μίντια που είναι κατά της κυβέρνησης και μπορούν ελεύθερα να πούν ό,τι θέλουν. Με βάση στοιχεία ή χωρίς στοιχεία. Υπάρχει αυτό. Το είπα. Αν δείτε τα εβδομαδιαία έντυπα, όλα είναι κατά της κυβέρνησης. Όλα. Και κατά του Προέδρου. Ανεξαιρέτως. Από τις ημερήσεις εφημερίδες έχουμε τουλάχιστον τρεις. Τρεις. Δύο είναι εντελώς κατά της κυβέρνησης και μία είναι πάνω κάτω αντικειμενική. Μπορείτε να τα αγοράσετε αυτά ε, τα έντυπα. Υπάρχουν. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα ε, περίπτωση της Βράνσκα Νόβινε πριν από 10 μέρες, μια τοπική εφημερίδα που είπε ότι τους έκλεισαν γιατί δεν τους στήριζε η κυβέρνηση. Επέκνα την κυβέρνηση, δεν είχαν χρήματα και τους κλείσαμε. Ζήτησα αναφορά και έκθεση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Ενημέρωσης και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι έγινε. Βεβαίω επικρίνει την κυβέρνηση αυτό το μέσο και μπράβο του, δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Το 2017 και μόνο έλαβε από την κυβέρνηση ακριβώς λόγω της ανεξάρτητης επιτροπής στο Υπουργείο Πολιτισμού που χρηματοδοτεί τα έργα, έλαβαν περισσότερα χρήματα από ότι την τελευταία πενταετία, από το 2008, μάλλον από το 2008 μέχρι το 2012 και το 17 και μόνο πήραν περισσότερα κονδύλια. Όταν έβγαλα αυτά τα στοιχεία, και να μην μιλάμε για αίσθηση που έχουμε και για αντίληψη για τα πράγματα, αλλά με στοιχεία. Όταν βγήκα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, τι είπανε η αντιπολίτευση, ότι εντάξει, αλλά άλλοι πήραν περισσότερα. Το πρώτο που είπαν ότι μας κλείσατε ε, γιατί δεν μας δώσατε λεφτά. Όταν αποδείχθηκε ότι τους δώσαμε και περισσότερο από ότι μέσα σε πέντε χρόνια στο παρελθόν, από το 2008 μέχρι το 2012, ήρθε το άλλο επιχείρημα, ναι, αλλά κάποιοι άλλοι πήραν παραπάνω. Πάντως είμαι πρόθυμη να συζητήσω αυτό το θέμα, να το κατανοήσω καλύτερα και να δω τι μπορούμε να κάνουμε, αν πραγματικά είναι ζήτημα. Ευχαριστώ. Minister, thank you. Ευχαριστούμε, κυρία Πρωθυπουργέ, ο Πρόεδρος. Και πάλι σας ευχαριστούμε. που απαντήσατε με τόση ευθύντα και ειλικρίνη σε αυτές τις ερωτήσεις. Ε, για μας βέβαια είναι κάτι ξεχωριστό τον έρχεται στην Επιτροπή μας μία πρωθυπουργός. Ε, θελήσατε κι εσείς να έρθετε και αυτό φαίνεται το πόσο φιλοευρωπαϊκός είναι ο προσανατολισμός σας. Ε, καλή τύχη στις μένες συνομιλίες με τον πρώτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύριο με τους επιτρόπους και καλή επιτυχία στην εκδήλωση για την Κοϊκοντίνα απόψε. Καλή τύχη για το έργο σας. Καλή τύχη για τη χώρα σας και θα σας βοηθήσουμε στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή.